Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Να σας γνωστοποιήσω ένα καλό νέο και ένα λιγότερο καλό. Πρώτα το καλό. Μετά από πολλές ανατροπές τελικά βρέθηκε συμφωνία για το ε, ντοσχε fc FC2 ενώ η προδρία δεν περίμενε να γίνει συμφωνία και δεν κατάφερε να γίνει συμφωνία στον τριμερή διάλογο στο Στρασβούργο στις 26 Οκτωβρίου. Το Κορεπέρ την επόμενη μέρα δέχτηκε τους όρους της συμφωνίας, η οποία επισήμω εγκρίθηκε στο Κορεπέρ στις 8 Νοεμβρίου, χθες. Το κείμενο λοιπόν θα αποτελέσει αντικείμενο στην ψηφοφορία της Ολομέλειας το Δεκέμβριο και θα τεθεί σε εφαρμογή ε, στις αρχές του 2018 να συγχαρώ τον Χωζέ Μανουέλ Φερνάντε, τον εισηγητή μα, ο οποίο όμω δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το πρωί. Θα ε, δεχθεί τα εγκόμια που θα τα απευθύνουμε. Το λιγότερο καλό νέο. Η συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου. Σήμερα στις 11.30 θα γίνει τριμερής διάλογος στο Συμβούλιο η Επιτροπή αμέσως ε, ανέλαβε μέσω του Επιτρόπου να μας ε, αποστείλει το έγγραφο με τις συμβαστικές προτάσεις και πραγματικά αυτό ε, το έπραξε ο Επιτροπός γιατί το λάβαμε το έγγραφο ήδη την Τρίτη το πρωί. Μετά από την ανάγνωση του Κοινοβουλίου, η διαπραγματευτική μας ομάδα δεν θεωρεί ότι είναι καλή βάση για συζητήσεις το έγγραφο αυτό. Διότι με την ενδιάμεση αναθεώρηση και έχοντα αποδεχτεί αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση έχουμε χάσει κάθε διαπραγματευτικό περιθώριο στα πλαίσια αυτού του πολυετούς ε, προγράμματος. Δεν ξεκινάει λοιπόν με τους καλύτερους ιονούς αυτή η συνδιαλλαγή, αλλά θα προχωρήσουμε. Χθε συνάντησα τον Επίτροπο μαζί με τον κύριο Μωρεσάν, τον Γενικό μας και ο Επίτροπος είπε ότι είναι απλώ μια πρώτη φάση στην όλη διαδικασία. Περιμένουμε λοιπόν και το επόμενο έγγραφο. Αυτό που υπονοείται εδώ και που μας ενδιαφέρει να τονίσουμε είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε το μέγιστο δυνατό περιθώριο ευελιξίας διότι μπορεί το 2018 να χρειαστεί να ε, αποδώσουμε στην Τουρκία 3 δις. Και αρχικά προβλεπόταν ο προπολογισμός της Ένωσης να δώσει το 1 δις και τα 2 δις ε, τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή μάθαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα δώσουν τίποτα και τα τρία δις θα πρέπει να τα βρούμε από τον προπολογισμό της Ένωσης. Αυτό μας φέρνει σε μια δύσκολη θέση, διότι μπορεί να αναρωτηθούμε αν το σχέδιο προπολογισμού ήταν έντιμο στο βαθμό που δεν αναφέρει ξεκάθαρα ε, αυτά που θα έπρεπε να αναλυθούν την επόμενη χρονιά. Πέραν αυτών, ελπίζουμε ότι στις 17 θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, είναι Παρασκευή, θα έχετε και τη μετακίνηση Στρασβούργο-Βρυξέλλες και θα πρέπει να το κάνετε για να λάβετε μέρο, θα πρέπει να το κάνουμε για να λάβουμε μέρος σε αυτή τη συνδιαλλαγή. Ελπίζουμε λοιπόν να οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά έχουμε και σοβαρές αμφιβολίες. τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Θα σα στηρίσουμε ενήμερου για την πρόοδο των συζητήσεών μας και νομίζω ότι σήμερα το πρωί ο τριμερής διάλογος θα είναι πολύ σύντομος, διότι το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει διαπραγματευτική εντολή και δεν είναι σε θέση να δείξει την απαραίτητη ευελιξία για να έρθει πιο κοντά στις δικές μας ε, ε, απόψεις. Και τώρα να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Περιμένουμε λίγα λεπτά, διότι ήταν προγραμματισμένες στις 9 ακριβώς. Σας παρακαλώ να σπρώξετε τις κάρτες σας στα ηλεκτρονικά μηχανήματα για να κάνουμε μία πρώτη δοκιμή. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Περιμένουμε ακόμα κάποιους. Εγώ ψήφισα. Bon, eh bien, της προφορίας. Με πολύ θετικό αποτέλεσμα, 16 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Και τώρα θα ψηφίσουμε για την έκθεση του Ντανιέλ Λεβιώτη για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αλμαβίβα. Τροπολογία 1 υπέρ. Θα έπρεπε να διευκρινίσω ότι είναι η πρώτη τροπολογία μαζί με την προφορική της τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 ψήφισαν άπαντες. Λείπουν τρεις. Δεν λειτουργεί το μηχανημά σας. Μπορέσατε να ψηφίσατε ή όχι, θα μας πείτε ε, τι ψηφίζετε. Κάποιος δεν ψήφισε, πέραστε τις ψηφοφορίες. 16 υπέρ, 3 κατά, μία εποχή. Κυρία Τομά, τι ψηφίσατε. 18 συνολικά, 18-3-1. Συγχαρητήρια στον κύριο Βιώτη. για την έκθεση Γκέγερ. Γκάγερ για την ακριβία. για την ε, ποινική δίωξη απάτριβων. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 2 καταπέπτει και η 14 το ίδιο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 μάλλον 7 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα οι αιτιολογικές σκέψεις. 1 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν παντες πέρας. 19-3. Κυρία Τωμά. Κατά. Α, υπέρ. 20. Η κυρία Διέ. Αποχή. 19-20 μάλλον 3-1. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκάγερ. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Γκάγερ Εάν όμω δεν υπάρχει αντίρρηση, να δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Κύριε Ούρελ, για αυτή τη μεταφορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν κατάλαβα καλά, θέλατε να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για όλε τι μεταφορέ. Λοιπόν, μεταφορά 19 είναι η μετάφραση στον προπολογισμό τη κινητοποίηση του Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, η οποία μόλι ψηφίστηκε πριν από 10 λεπτά από την Επιτροπή σα. Μια καθιερωμένη μεταφορά από το αποθεματικό στη βασική δημοσιονομική γραμμή. Η μεταφορά 21 αφορά την κινητοποίηση 18 εκατομμύρια ανάληψη χρώσεων και χρήση 26,5 εκατομμύρια από άλλη δημοσιονομική γραμμή και τα δύο με σκοπό να ενισχύσουν την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Να θυμίσω ότι πριν το καλοκαίρι η Επιτροπή αυτή είχε ψηφίσει και εγκρίνει τη μεταφορά υπαριθμών 9. Είχαμε μεταφέρει 85 εκατομμύρια από τον προπολογισμό CFSP στην ε, ε, διευκόλυνση για την ε, κάλυψη των προσφύγων στην Τουρκία. Και σα είχα πει ότι θα κοιτάξουμε τον προπολογισμό του CFSP αργότερα μέσα στη χρονιά, πράγμα που μόλι κάναμε. Τώρα εντοπίσαμε τι ανάγκε που προέκυψαν και μπορέσαμε να δούμε πού χρειάζεται νέα χρήση ποσών. Μέσω λοιπόν από τον επανασχεδιασμό αυτή τη στρατηγικής χρειαστήκαμε τα 18 εκατομμύρια από το αποθεματικό για τι επίγουσε ανάγκες. Προς ενημέρωση των μελών να πω ότι μετά και εφόσον εγκριθεί αυτή η μεταφορά για την υπόλοιπη χρονιά θα έχουμε 61,7 εκατομμύρια στο αποθεματικό για τις επίγουσες ανάγκες. Κατά την άποψή μας είναι ε, περισσότερο από ό,τι χρειάζεται για να καλύψουμε τις προβλεπόμενες ανάγκες. Τώρα η μεταφορά 23. έτοιμα για να χρησιμοποιήσουμε από την γραμμή για τις αλληλευτικές συμφωνίες προς την ε, λειτουργική γραμμή του προπολογισμού μετά τις διμερείς συμφωνίες αλληλευτικής εταιρικής σχέσης για τη Μαυρικτανία, το Μαυρίκιο, τις Ειχέλες και το Κυριμπάτι. Από νομικής σκοπιάς αυτό πρέπει να έχει εγκριθεί στις 15 Νοεμβρίου, οπότε θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάγερ, ο οποίος το προέβλεψε στην ημερήσια διάταξη αυτή τη ε, ε, Επιτροπή εγκαίρω για να γίνει αυτή η ψηφοφορία όπω πρέπει για την 24 πρόταση της Επιτροπής να μεταφερθεί κονδύλι που έχει γίνει διαθέσιμο από, το, από τη μισθολογική γραμμή της Επιτροπής για να ενισχυθούν οι δαπάνες IT και να καλύψουμε κάποιες σχετικά επίγουσες ανάγκες που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή μετατροπή και να μπορέσει η Επιτροπή να προετοιμαστεί για το ψηφιακό εργασιακό χώρο του μέλλοντος. Θα σας ζητούσα λοιπόν για να ξεκινήσει η αντικατάσταση του λογιστικού συστήματος ΑΜΠΑΚ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει φτάσει στο τέλο τη ζωή του να εγκριθεί αυτό το κονδύλι. Ο λόγο που το κονδύλι αυτό διατέθηκε από τη μισθολογική γραμμή είναι γιατί δεν μπορέσαμε να προσλάβουμε όσο εγκαίρω πιστεύαμε, γιατί δεν υπήρχαν υποψήφοι από τον κατάλογο επιτυχόντων για την ε, μεταφορά 28 ενίσχυση, να ε, ενισχύσουμε το τελωνιακό πρόγραμμα κατά 7 εκατομμύρια περίπου, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει τις νομικές υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Κώδικα και ορίσαμε κάποιες ε, νέες ανάγκες, κυρίως για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Ουσιών Και επίσης πήραμε και από τον προπολογισμό ΕΑΖΑ και από το Γραφείο ε, Δημοσίευσεων. Επίσης 29 πρόταση να ενισχύσουμε το πρόγραμμα τροφίμων και ζωοτροφών κατά 2,7 εκατομμύρια και σε πληρωμές και σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Αυτό για να βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες της γρήπης των πουλερικών. Και επίσης μεταφορές και επίσης για δαπάνες από το εργαλείο κάλυψης επιγουσών αναγκών και το μηχανισμό προστασίας. Τελευταία μεταφορά που θα πρέπει να εγκρίνεται σήμερα είναι η περίθμον 30, κάτι που επανέρχεται κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο τέλος της χρονιάς κλασικά να μεταφερθεί από τη δαπάνη διοικητική στήριξη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλε γραμμέ, στι λειτουργικέ γραμμέ του προπολογισμού, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, προ όφελο των διαφόρων προγραμμάτων, κυρίω για την ενίσχυση των λειτουργικών γραμμών του ορίζοντα 2020 και σε μικρότερο βαθμό του ΙΤΕΡΣΕΦ και του Κόσμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επομένω υπάρχει ανάγκη κονδυλίων για την τροπολογία 30. Κύριος Γκάιερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μου σκοπιά, η πλειονότητα αυτών των μεταφορών πιστώσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να προκαλεί πρόβλημα. Για μια ιδιο θα ήθελα μια αναβολή, διότι έχω κάποιες ανάγκες διευκρινήσεων ακόμα. Επομένως, για τη 19 όντως την έχουμε ήδη ψηφίσει, έκθεση διότι θα ήταν περίεργο να την εγκρίνουμε πολιτικά και μετά να μην δώσουμε τα χρημα... τη χρηματοδότηση. Τώρα, για την 21 ωστόσο είναι κάπως πρόβλημα, διότι είχαμε λάβει ήδη από το κονδύλιο αυτό με την DEC 7, με τη μεταφορά 7 δηλαδή, χρήματα, διότι είχε τότε αιτιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειαζόταν τα κονδύλια αυτά. Τώρα όμως τα χρειάζεται και πάει να κάνει εκ νέου επανακατανομή. Εγώ δεν λέω ότι αυτό αποκλείεται καταρχήν αλλά δεν δείχνει έτσι, πολύ πιστική διαχείριση του προπολογισμού. Ας κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς έχει γίνει, αφού άλλωστε όπως είπε και ο πρόεδρος μας Αρτουή, μίλησε για την παράταση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Αυτά όλα μπαίνουν σε μια συνολικότερη εικόνα, όπου μπαίνουν όλα τα εργαλεία της εξωτερικής πολιτικής και τα οποία έχουμε ελέγξει για να δούμε τι μπορεί ω κονδύλιο δηλαδή να απελευθερωθεί από κάποιο από αυτά για την διευκόλυνση των προσφύγων στην Τουρκία. Εγώ θεωρώ ότι πολιτικά υπάρχει λόγος να αξιολογηθεί ξανά, να δούμε δηλαδή όλο αυτό το patchwork πώς ε, θα διορθωθεί. 23-24 χωρίς πρόβλημα. 28 θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρώτα χαίρομαι που ε, εισπράττονται τέλη εισφορές και έτσι μπορούν να αλαφρώσουν κάπως τον προϋπολογισμό από τον οργανισμό αυτό δηλαδή εισπράττονται εισφορές. Αλλά είναι μια υπόθεση που την παρακολουθώ από τότε που μου ορίσατε εισηγητή για τους οργανισμούς, για τους προϋπολογισμούς των οργανισμών Όπου δηλαδή μπορεί να αυξηθούν οι εισφορές χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα, είναι σωστό να εισπράττονται και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Να δηλαδή, επιβαρύνονται δηλαδή, δηλαδή με τις εισφορές αυτές οι πελάτες των οργανισμών και να ελαφρώνεται ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Ωστόσο υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο στα μάτια μου πότε ενημερώνονται οι οργανισμοί για την μεταφορά πιστώσεων. Διότι η ΕΑΣΑ κάνει μάλιστα ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα, το οποίο έχουμε εγκρίνει και εμείς, και από όσο ξέρω, τουλάχιστον από τα τελευταία νέα σήμερα το πρωί, είναι ότι χρειάζεται η ΕΑΣΑ τα χρήματα αυτά για το πιλωτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό θα έλεγα να ανασταλεί, να αναβληθεί μάλλον η 28. Το ίδιο για την 30. Θέλω να, να, τα, έχω, να τα πω αυτά πάντως για να τα ακούσουν οι συναδελφοί μου. Τώρα η ΙΤΑ, όπως είπα πριν, για την 18, μεταφορά πιστώσεως 18, είπε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται χρήματα. Τώρα πάει να τη χρηματοδοτήσει. Εάν τελικώ αποδειχτεί ότι μέχρι το τέλο του έτου δεν τα χρειάζεται ο οργανισμό αυτό τα χρήματα αυτά, τότε αυτά θα επιστραφούν στα ταμεία των χωρών μελών. Αλλιώ τα πλέον ο οργανισμό από μόνο του. Αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση η Κομισιόν. Το καταλαβαίνω απολύτω. Και υπάρχει βέβαια ε, ο καυγά για το πάπλωμα. Ή τραβάει ο ένα από εδώ, ή τραβάει ο άλλο από εδώ. Πότε κρυώνει το, κρυώνουν τα πόδια, πότε κρυώνουν οι ώμοι και ο λαιμό. Τι να κάνουμε. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εντολή των χωρών μελών ε, να εφαρμόζει πολιτικές και να τις χρηματοδοτεί. Όπου λοιπόν η μετακίνηση αυτή των δημοσιονομικών κονδυλίων αρχίζει και φαίνεται λίγο παράδοξη, τότε θα πρέπει να καθόμαστε να τα συζητούμε, διότι αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία άλλωστε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εναντί των χωρών μελών για να τους εξηγήσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τον προπολογισμό δεν είναι απαραίτητο καλύτερο για την εφαρμογή των πολιτικών που οι ίδιες έχουν εγκρίνει. Ευχαριστώ ε, κύριε Σιγητά. Γενική Σιγητά του Άρα θέλετε για 21 και 28 αναβολή. Μάλιστα. Η κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα μου εξήγησαν ότι για τα ακίνητα και αναφέρομαι στο 24 και ιδίω για αντιπροσωπείες που βρίσκονται σε δύσκολες περιοχές υπάρχουν έξτρα ανάγκες ασφαλείας. Χρειάζεται πρόσθετο, χρειάζονται πρόσθετο εξοπλισμό πολλά από τα κτίρια αυτά, ώστε να προστατεύονται κατάλληλα οι, ε, οι εργαζόμενοι. Δεύτερο, για τους οργανισμούς. Έχω μια προσθήκη εδώ, αγαπητέ Γιάννη Γκάιερ, σε ό,τι αφορά την αύξηση των εισφορών, διότι είχαμε πει από την αρχή ότι ιδίω οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται υπερβολικά. Δηλαδή, τελικώς, να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητήσουν αδειοδότηση για τις διάφορες χημικές συνθέσεις που ε, παράγουν, που έχουν στην παραγωγή τους, δηλαδή να επιβαρύνονται έξτρα με υψηλές εισφορές και τέλη. Και αυτό ιδίως για χώρες οι οποίες μάλιστα αντιμετωπίζουν οικονομικές ε, δυσκολίες. Ακόμα βέβαια αυτό ισχύει και για όλες τις χώρες. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν μπορεί να γίνει χωρίς αύξηση των τελών, διότι εδώ εμείς κάνουμε μεταφορά πιστώσεως. Θα ήθελα ή δυνατόν να αποφευθεί λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα κάπως περισσότερες εξηγήσεις. Να μην λέμε ότι εμείς κάνουμε εδώ μεταφορές πιστώσεων στον υπολογισμό, οι οποίες ωστόσο οδηγούν στο να αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να καταβάλουν υψηλότερες εισφορές στους οργανισμούς της Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ανάλυση που έκανε και με την οποία συμφώνω έχω κάποιες ερωτήσεις τώρα για τη μεταφορά πιστώσεων 21. Είναι λίγο περίεργο ότι τον Ιούνιο παίρνουμε χρήματα από τη διευκόλυνση για την Τουρκία για να τα δώσουμε αλλού και τώρα παίρνουμε από αλλού για να τα δώσουμε εκεί, στη διευκόλυνση για την Τουρκία. Ε, θα ήθελα να μάθω τι γίνεται, διότι δεν είχα φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, μία ερώτηση για την 4. Το σύστημα υπολογισμών ABAC. Το συνολικό κόστος δεν είναι σαφές για μένα, πάντως δεν βρήκα κάποιο συγκεκριμένο αριθμό. Το ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαμε να λάβουμε κάποια στιγμή ένα έγγραφο, το οποίο να περιγράφει συγκεκριμένα τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες μέχρι το 2022 για τον εξυγχρονισμό του συστήματος. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο και για τις ε, παραπέρα εργασίες μας, διότι το Κοινοβούλιο παρακολουθεί την εξέλιξη του συστήματος αυτού. Και τώρα, μια στιγμή, για την 28, για τον ε, τελωνιακό κώδικα. Εδώ εξηγείται καλά ότι οι χώρες μέλη συμφώνησαν το, η αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου να ανασταλεί μέχρι το 2023, αλλά πώς ζητάτε τώρα να, να θεωρηθεί το προηγούμενο. Θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα. Μήπως και αυτό πρέπει να το θέσουμε ως πρόβλημα στο Συμβούλιο για να επιτευχθεί κάποια καλύτερη λύση. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Πρώτα εσείς κύριε Γιουρέλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθήστε να απαντήσετε παρακαλώ στις ερωτήσεις που σας έγιναν. Ευχαριστώ από την πλευρά μας μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση του κυρίου Γκάιερ να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την ΤΕΚ 28. Επίσης σημείωσα ότι υπήρξαν και πολλές ερωτήσεις ως προς αυτό. Οπότε μπορούμε να επανέλθουμε απαντώντας τις ερωτήσεις ε, και από την κυρία Χολμάιερ και από την κυρία Γκρέσλε. Όσον αφορά την ΤΕΚ 21, αυτό είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί χρειαζόμαστε τα κονδύλια αυτά για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις αποστολές ε, CFSP, οι οποίες προβλέπεται να πληρωθούν κατά τις ερχόμενες εβδομάδες. Και είναι εδώ ο συνάδελφος, ο τμήματάρχης, ο Κριστιό Μινιέ, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να δώσει περισσότερες πληροφορίες ως προς αυτό, αλλά για να σας εξηγήσω μία ακόμη φορά την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποια ε, ασάφεια ως προς αυτό. Πριν από το καλοκαίρι σας είχαμε προτείνει και είχατε συμφωνήσει να ψηφίσουμε τα 85 εκατομμύρια από τη δημοσιονομική γραμμή, από τη γραμμή προπολογισμού του CFSP για τους πρόσφυγες ε, στην Τουρκία. Ήταν κατεπήγον, ε, είχαν εντοπιστεί ανάγκες για τα σχολεία, τα παιδιά, για τους πρόσφυγες του Σύριου της Τουρκίας και είχαμε πει ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εξηγήσει ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπρόσθετες ανάγκες, τι ανάγκες θα υπάρξουν για τον προϋπολογισμό CFSP για αυτή τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ νωρί για να έχουμε μία σαφή εικόνα. Εν τω μεταξύ όμως έχουν περάσει τέσσερις μήνες, η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει, κάποιες νέες αποστολές έχουν αποφασιστεί και τώρα είναι πλέον σαφές ότι ο προϋπολογισμός της FSP ε, χρειάζεται να ενισχυθεί. Όμως το γεγονός ότι αναβάλαμε την απόφαση αυτή ε, για τέσσερις μήνες σήμαινε ότι μπορέσαμε να τα καλύψουμε μέσω επαναδιάθεσης και μέσω ανακτήσεων ποσών από προηγούμενες ε, αποστολές. Άρα μόνο 18 εκατομμύρια ε, της ε, κατεπίγουσας, ε, των κατεπηγόντων ποσών, της κατεπίγουσας βοήθειας χρειάζεται. Καταλαβαίνω βέβαια τους δισταγμούς σας και τους ενδιασμούς σας. Πρέπει να σας πω τις ίδιες επιφυλάξεις άκουσα και από το Συμβούλιο. Βεβαίως σημειώνουμε αυτήν την κριτική και θα τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη για το μέλλον. Γιατί δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος ε, να ε, προχωρούμε. Πάντως θα ήθελα να σας ζητήσω αν είναι δυνατόν ε, να κάνουμε την ψηφοφορία σήμερα και ίσως ο συνάδελφος για ένα-δύο λεπτά να σας εξηγήσει λίγο περισσότερα. Ευχαριστώ. Για την 21 λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μακάλιστερ ε, συμμετέχει επίσης. Ε, πριν από ένα μήνα είχαμε αποφασίσει, είχαμε πει, είχαμε διαπιστώσει ότι μας λείπουν 50 εκατομμύρια. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Ρέιλ ότι πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, είναι πλέον κατεπίγουσα η κατάσταση. Μπορείτε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το κατεπήγον της κατάστασης, τρεις μεγάλες αποστολές σε CFSP πρέπει να ανανεώσουμε από σήμερα μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, Γεωργία, Λιβύη και Ουκρανία. Αυτές τις τρεις έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει με προκαταβο... με... αναμένοντας την ενίσχυση του της σημερινή ε, της αποστολής στο Ιράκ η οποία αποφασίστηκε πριν από δύο εβδομάδες από το Συμβούλιο και η οποία αυτή τη στιγμή έχει ήδη δρομολογηθεί. Πρόκειται για μια νέα αποστολή που δεν προβλεπόταν στην αρχή της χρονιάς είναι ένας παράγων ε, επί του οποίου δεν είχαμε ακόμη πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά στοιχεία, δεν ξέραμε ακριβώς τι θα γίνει. Τώρα το γνωρίζουμε καλύτερα γιατί μέχρι το τέλος ε, του μήνα πρέπει να αποφασίσουμε και πριν επειδή θα πρέπει να δώσουμε γύρω στα 80 εκατομμύρια μας, ε, χρειαζόμαστε ακόμη κάποιες πιστώσεις, έχουμε κάνει κάποιες ανακτήσεις ποσών, χρειαζόμαστε όμως τα ποσά αυτά γιατί υπάρχουν εκατοντάδες άτομα που ε, επανδρώνουν αυτές τις αποστολές και χρειαζόμαστε τα ποσά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρέλ, το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Υπήρξαν κάποιε ερωτήσει ακόμη όσον αφορά τι 10, 24 και 30. Όσον αφορά την 24, η κυρία Χολμάιερ έκανε μία ερώτηση ε, σε σχέση με τις ανησυχίες που υπάρχουν για την ασφάλεια των κτηρίων, να σας καθησυχάσω ότι έχουμε κάνει μια εκτίμηση της γραμμής προπολογισμού. Ε, είναι χαμηλότερη η αξιοποίηση φέτος από την αναμενόμενη και ο λόγος δεν είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, αλλά ε, επειδή έχει αυξηθεί η αξία του ε, ευρώ σε σχέση με τη στιγμή που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός. Πρέπει να πω λοιπόν ότι αυτό είναι μια καλή εξέλιξη λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε, τη σημειώνω περισσότερες πληροφορίες ε, για το πρόγραμμα ABAC. Πιστεύω ότι μπορώ να σας τις παρέχω αυτές. Μία ακόμη ερώτηση για το, από τον κύριο Γκάιερ για την DEC 30. Αυτή είναι η τελευταία νομίζω σε σχέση με την ΙΤΕΡ. Καταλαβαίνω απολύτως ότι δεν είναι πάρα πολύ διαφανής ε, η παρουσίαση. Αυτό που συμβαίνει όμως ε, είναι ότι ουσιαστικά ένα ταυτόσιμο ποσό 1,1 εκατομμυρίου ε, από μία γραμμή διοικητική ε, το μεταφέρουμε σε μία επιχειρησιακή γραμμή. Και όπως ξέρετε, για να γίνει αυτή η μεταφορά δεν μπορεί ε, να την αποφασίσουμε μόνοι μας. Πρέπει η αρχή του προπολογισμού να ε, συμφωνήσει και εκείνη, να μην υπάρχει δηλαδή ούτε υποαξιοποίηση ούτε υπερβολική εκτέλεση. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια απλή μεταφορά 1,1 εκατομμυρίων από διοικητική γραμμή σε επιχειρησιακή γραμμή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέλ. Ε, έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Κύριε Γκρέσλε. Ερώτηση 28 για το σύστημα λογισμικής, λογισμικού, συγγνώμη, το ABAC. Για την, 28 ε, δεν ε, υπάρχει πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα. μπορώ να σας απαντήσω κι εγώ. Ε, έχετε το λόγο αν θέλετε να πείτε κάτι. Ήθελα να επανέλθω όσον αφορά το ερώτημα αυτό της κυρίας Γκρέσλες με γενέστερο στάδιο. μπορώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες γραπτός όμως, αν μπορείτε να το δεχτείτε αυτό. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Γκρέσλε. Πολύ ωραία. Κύριε Σιγητά. Ε, κύριε Ερέλ, μπορώ να κατανοήσω την επιχειρηματολογία που προβάλλεται για το ΔΕΚ 21. Δεν θα κρατήσει η παρούσα Επιτροπή χρήματα τα οποία ενδέχεται να χρειάζονται αλλού Θεωρώ πάντως ότι πρέπει να ε, προειδοποιήσουμε το Συμβούλιο. Δεχόμαστε την διαχείριση αυτή, διότι το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση ε, να διαθέσει νοπό χρήμα για να αντιμετωπίσει να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις ασφαλείας οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν το 2013 όταν άρχισε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και είπαμε 3 δισεκατομμύρια για την Τουρκία, από τα οποία το ένα θα διατίθεται από τον ε, κοινοτικό προπολογισμό και τα δύο από τι χώρε μέλη. Τι θα γίνει τώρα εάν ισχύσουν οι γνώμε ορισμένων χωρών μελών, η επόμενη δόση των 3 δισεκατομμυρίων να διατεθεί ολοσχερό από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εγώ δεν έχω διάθεση να συγκρίνω κάτι τέτοιο τότε θα υποβάλω τροποποιημένη πρόταση στην ε, Επιτροπή Προϋπολισμών να εγκρίνει όλες τις προτινόμενες μεταφορές πιστώσεων με εξαίρεση την υπαριθμών 28. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Πράγματι υπάρχει επίγον και υπάρχει μια παράδοξη κατάσταση διότι υπάρχει υποεκτέλεση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑ, όμως τούτη τη χρονιά έχει ανατραπεί η κατάσταση και τα κονδύλια τα οποία έχουν αφαιρεθεί από την ΚΕΠΑ την θέτουν σε κίνδυνο διότι τώρα είναι ελληματική. Κύριε Σιγητά, μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις μεταφορές με εξαίρεση την 28, η οποία θα ε, γίνει αντικείμενο νέας εκθέσεως. Λοιπόν, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Ψηφίσατε. Τέλος. Κυρία Τωμά, ψηφίσατε υπέρ, κυρία Βιού επίσης. Άρα, 23 ψήφοι υπέρ, Τρεις κατά και καμιά αποχή. Ο κύριος Τάραντ τώρα για τις μεταφορές για τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Έχει το λόγο κύριε Ισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη εισαγωγή που θα φανεί ότι δεν ταιριάζει στην ε, παρούσα συζήτηση, αλλά προ 28 ετών έπεσε το τείχος του Βερολίνου και αυτό επέτρεψε στις κυρίες Βάιντερ, Σούλη, στον κύριο Σεχόφσκι, στον κύριο Μάρκα, σε μένα να συμμετάσχουμε στην ε, διακεκριμένη αυτή συντροφιά, όπως και η κυρία Γκρέσλε και άλλοι. Ήταν λοιπόν σημαντικό γεγονός στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενότητας και των αξιών της. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε εδώ για να δεχόμαστε κάθε είδους πρακτική που έχουν αναπτύξει οι παλαιές χωρίς μέλη. Και ιδίως για μια συγκεκριμένη μεταφορά πιστώσεως που ενδιαφέρει και τους φίλους της Επιτροπής Περιφερειών για την 1η Δεκεμβρίου του 2017 μιλώ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν φορετικές απόψεις, αλλά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη δική μου αντίληψη για το θέμα. Ο, το θεσμικό όργανο είχε ένα προϋπολογισμό στην αρχή του χρόνου με τον οποίο θα έπρεπε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες πολιτικών ομάδων και ούτω καθεξής. Ε, διαφωνώ να μεταφέρονται κάποιες δαπάνες για project επικοινωνίας, διότι τα θεσμικά μας όργανα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν σε τέτοια κλίμακα που κανένα σχέδιο μας ακούει. Ξέρω ότι συμφωνείτε, ότι, συγγνώμη, ότι διαφωνείτε κυρία Χολμάιερ. Αλλά να ε, να σας εξηγήσω γιατί το σκέπτομαι αυτό. Ο προϋπολογισμός όταν αντιμετωπίσαμε την δημοσιονομική κρίση, είχαμε συμφωνήσει να γίνουν κάποιες περικοπές, 5% στο προσωπικό για 5 χρόνια και διάφορα Και διαπιστώνουμε ακόμη ότι υπάρχουν πόροι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις, δηλαδή πόροι τους οποίους δεν χρησιμοποιούμε. Και ίσως υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά αυτά παρά να διατεθούν για επικοινωνία και να ανοίγουν γραφεία εκπροσώπησης και να προσλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι θα στέλνουν tweet και είμαι σίγουρος ότι το Twitter ως, ως φαινόμενο των κοινωνικών μέσων προωθεί στην ουσία τον αναλφαβητισμό, την ακατανοησία, δεν κάνει καλά πράγματα δηλαδή, να μην σας πω καθόλου για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έτσι, και τον λογαριασμό Twitter που διαθέτει, Κατά τη γνώμη μου λοιπόν η Επιτροπή Περιφερειών μπορεί μια χαρά να τα καταφέρει και χωρίς τη μεταφορά πιστώσεως και τίποτα κακό δεν θα πάθει. Αυτή πάντως είναι η προσωπική μου άποψη. Και σας ευχαριστώ που την ακούσατε και ας ψηφίσουμε. Αλλά οι άλλες πιστώσεις, οι άλλες μεταφορές δηλαδή δεν είναι προβληματικές στα μάτια μου. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. παρεμβάσεις. Κυρία Χολμάιερ, πολύ σύντομα. Έχοντας αποφασίσει η Επιτροπή Περιφερειών, προβλέπεται στον προϋπολογισμό, τους επικρίνουμε συχνά ότι δεν κάνουν καλή επικοινωνία. Και τώρα που κάνουν, πάνε να κάνουν μια προσπάθεια, και αυτό δεν ισχύει μονάχα για το Twitter, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα για το Twitter, αλλά δεν πρόκειται μόνο για το Twitter. Οι αποφάσει των οργάνων τη Επιτροπή Περιφερειών δεν πρόκειται να ανατρέψουν και δραματικά τον προπολογισμό. Οπότε ίσω δεν θα έπρεπε να του ε, το απαγορεύσουμε. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί κανείς. Καλώς. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την μεταφορά για την Επιτροπή Περιφερειών ΔΕΚ 1 2017. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε. Κυρία Τωμά, ψηφίσατε υπέρ. Εσείς, κυρία Βιέ, επίση. Άρα, 18 ψήφοι υπέρ, 6 κατά και μια αποχή. Ο εισηγητή μα δήλωσε ότι οι υπόλοιπε αιτήσει μεταφορών πιστώσεων δεν ε, είναι προβληματικές ε, στα μάτια του και ότι μπορεί να συστήσει έγκριση. Εάν δεν υπάρχει καμιά ένσταση, εγώ θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Το λόγο λαμβάνει τώρα η κυρία Μόνικα Χολμάιερ για να αναπτύξει ένα θέμα σχετικό με την Φιλανδία. Έχει ζητήσει περισσότερες προφορίες, τις οποίες θα αναπτύξει τώρα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, πρόκειται πάλι για την κτηριακή πολιτική και το έργο της ΕΚΑ, Οργανισμός που έχει την έδρα του στο Ελσίνκι και που έχει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2019. Πρέπει λοιπόν να συζητηθεί εάν θα παραμείνει ο οργανισμός αυτός στο ίδιο κτίριο ή εάν θα μετακομίσει. Έχει ξεκινήσει μια πλήρη διαδικασία με επαφές με πάνω από 100 εταιρείες ε, με σιτών, ακινήτων κλπ, με προκηρύξεις και εν τέλει ο οργανισμός αυτός έχει βρει ένα νέο κτίριο κοντά στο παλαιό κτίριο. Η τελευταία ανακαίνιση του παλαιού κτιρίου έγινε το 1980. Επομένω είναι απολύτω αναγκαίο να ανακαινιστεί εκ βάθρων, κάτι που θα σημάνει βέβαια δύσκολε και ταπανηρέ εργασίε. Και θα πρέπει βέβαια να εγκαταλείψουν το κτίριο για δύο χρόνια και μετά να επανακάμψουν. Έτσι λοιπόν ο, παραγωγισμός ΕΚΑ θεωρώ δικαίως αποφάσισε να αναζητήσει νέα εγκατάσταση, νέο κτίριο. Το οποίο νέο κτίριο βρίσκεται στο Business District του Ελσίνκη. Είναι δύο ξεχωριστά κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους και το νέο συμβόλαιο θα πρέπει να είναι από το 2020 έως 2030 με επιλογή παράτασης για μια πενταετία ακόμα το κτίριο είναι κατασκευή 2019, δηλαδή δεν καν έτοιμο ακόμη, άρα είναι απολύτως καινούριο, ε, μπορεί επομένως να προσαρμοστεί απολύτως στις ανάγκες του οργανισμού ΕΚΑ ή CHHA δηλαδή. Το συνολικό εμβαδόν του είναι 18.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το παλαιό κτίριο ήταν 24.000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά ήταν ε, ακατάλληλη κατανομή των χώρων γραφείων, άρα δεν εξυπηρετούσε. Ο οργανισμός λοιπόν ΕΚΑ έχει κάνει συστηματική εργασία το κόστος συνολικά. Τώρα παίρνω το ετήσιο κόστος μαζί με, όλα τα, με όλο το κόστος θα είναι της τάξης του, των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για το παλιό φτύριο ήταν 8,9 εκατομμύρια. Επομένως, πάλι κάπως εξοικονομούμε. Και εάν εξοικονομούμε και χρήματα, τότε μάλλον θα πρέπει να είμαστε υπέρ. Έχω πάντως την πρόταση, θα δούμε αν συμφωνεί η Επιτροπή Προϋπολογισμών, ο Πρόεδρος και εγώ να απευθύνουμε ερωτήσεις στον οργανισμό ΕΚΑ ή σύσταση αν θέλετε δεν υπάρχει δυνατότητα καταγγελία τη συμβάσεω. Δηλαδή, εάν φύγει ο οργανισμός ΕΚΑ μέσα στην δεκαετία, θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει κατά 100% το μίστομα μέχρι τέλους της συμβάσεω. Γι' αυτό κάνω τη σύσταση πρώτον να μπορεί να αναζητηθεί υπομισθωτή και δεύτερο να υπάρχει μια φθήνουσα δόση, δηλαδή όσο πλησιάζουμε στο τέλο ε, του μισθωτήριου συμβολέου ε, και αν εν πάση περιπτώσει ο εκμισθωτής έχει δύο χρόνια να βρει κάποιον ε, καινούριο μισθωτή να μην εισπράττει το 80% του μισθώματος. Δεύτερο, δεύτερη σύσταση, εάν γίνει αγορά, διότι υπάρχει και η επιλογή της αγοράς. Θα πρέπει πρώτα να ε, βουλιδοσκοπηθεί η αγορά, εάν δηλαδή η τιμή που θα προτείνει ο εκμισθωτής για αγορά του ακινήτου θα ανταποκρίνεται στις τιμές που ισχύουν στην αγορά. Αυτό ούτως ή άλλως θεωρώ ότι προκύπτει και ως υποχρέωση από τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτά λοιπόν, δηλαδή προτείνω έγκριση της μεταφοράς και αποστολή της επιστολής. Ευχαριστούμε κυρία Χολμάγερ για αυτήν την τόσο ξεκάθαρη και κρυστάλλινα ε, διάφανη επεξήγηση που μας δώσατε για όσα προτείνονται για αυτό το έργο. Κύριε Τάραν, ευχαριστώ. Απλώς να ενημερώσω εσάς και την εισηγήτρια ότι οι Φινλανδοί ε, είχαν ε, μετατρέψει την αμερικανική εκδοχή του Μονόπολη και την είχαν φέρει σε εμά στην Εστονία. Και το πιο ακριβό ήταν ε, όποιο κτίριο ανήκε στο business district του Χελσίνκη. Του Ελσίνκη. Uh, uh, uh, ναι, αλλά θα μπορούσαμε να αγοράζουμε και στις φθηνότερες περιοχές όπου η τιμή τους ε, θα ανέρθει αντί να πηγαίνουμε κατευθείαν στα ακριβά. Voilà une contribution au débat. Φοβερή συμβολή στη συζήτηση. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι φτηνότερα. Το ανάποδο ενός πλειοδοτικού διαγωνισμού. Πάντως, επειδή δεν εδώ ο κύριος Γκάγερ και γιατί μιλάμε για την πολιτική περιοργανισμών, θα έλεγα να περάσουμε στην ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη σύσταση της Μόνικα Χολμάγερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Κυρία Τομά, ψηφίσατε υπέρ. Κυρία Βία, επίσης. 24 ψήφοι υπέρ. 23, 23. Με συγχωρείτε. Λειτουργήσε. Επιτέλους. Ωραία λοιπόν. 23, 1 και μία αποχή. Για την πολιτική κτηρίων δεν έχουμε νέες πληροφορίες μόνικα. Ωραία λοιπόν. Θα ολοκληρώ... Ολοκληρώσαμε μάλλον με τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Και τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας Ράσβαν Πόπα για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για μία ε, κινητοποίηση στη Φινλανδία. Στις 12 Ιουλίου φέτος ε, η Φιλανδία έκανε αίτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από την απόλυση 160 ε, υπαλλήλων στο δυτικό τμήμα της χώρας. Το 2016 άρχισε η Φιλανδία να προσφέρει προ... Ε, εξατομικευμένες υπηρεσίες ε, για όσους είχαν απολυθεί, όπως για παράδειγμα καθοδήγηση για τη σταδιοδρομία, την βοήθεια σαν νεοφυείς επιχειρήσεις, κάτι το οποίο, το οποίο στήχιζε 2.499.360 ευρώ από το 76% των απολυθέντων είναι γυναίκες. Υπάρχει ένα θόρυβο στην αίθουσα που δεν ε, βοηθά κανέναν ε, εσείς εκπροσωπείτε τον κύριο Νεγκρέσκου που πήρε θέση στην κυβέρνηση και δεν σας διευκολύνει όλη αυτή η φασαρία που υπάρχει στην αίθουσα. Παρακαλώ λοιπόν να αποχωρήσετε ήσυχα. Καλημέρα σας κιόλα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, όπω έλεγα, αυτές οι υπηρεσίε θα στοιχήσουν 2.499.360 ευρώ στο ταμείο αυτό για 1.500 ε, ε, απολυθέντες, εκ των οποίων 76% είναι γυναίκες. Κάτι, ε, ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση είναι τα διαδικτυακά καταστήματα κυρίως αυτά εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, γιατί είναι το 90% όλων των ε, πολίσεων που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο. Αυτό θα πρέπει να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα όσον αφορά τα νέα προγράμματα ψηφιοποίησης, όχι μόνο στον τομέα του λιανικού εμπορίου, αλλά και σε άλλους τομείς. Η αίτηση λοιπόν έχει σκοπό να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους ε, να βρουν μια καινούρια δουλειά ή να ξεκινήσουν μια νέα ε, επιχείρηση, όμως ε, ο μέσος όρος είναι από τους χαμηλότερους 1.600 ευρώ κατά κεφαλήν. Γι' αυτό ακριβώς ζητώ την άμεση κινητοποίηση του ποσού αυτού που ανέφερα προηγουμένως που θα βοηθήσει αυτούς 1500 εργαζομένους ε, μέχρι τις 12 Ιουλίου ε, του 2019. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ποιο θα ήθελε να πάρει το λόγο προ αυτό. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές θα ανακύψει γιατί πάρα πολλοί φορείς ε, μεγάλων ε, καταστημάτων ε, υπεραγορών βρίσκονται σε κατάσταση που είναι έτοιμα να κλείσουν, να απολύουν ταμείες, ε, οι μεγάλες αλυσίδες διανομής ε, θα πληγούν πάρα πολύ από τις πωλήσει στο διαδίκτυο και αυτό πραγματικά θέτει ένα αμφιβόλο γενικότερα αυτή τη λογική της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, να, υπάρξουν όλο και περισσότερες αιτήσει στο ταμείο αυτό, για ενεργοποίηση του ταμείου αυτού στα επόμενα έτη. Οπότε το δικό σας συμπέρασμα βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση υπέρ της έγκρισης αυτής ε, της αίτησης. Ε, η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών είναι 16 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα, 20 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στην Επιτροπή μας και τέλη Νοεμβρίου, στη Μήνη Ολομέλεια εδώ στις Βρυξέλλες, θα γίνει η ψηφοφορία. Τώρα το λόγο έχει η Μαρή Πιέρ Βιέ, η οποία πρώτη φορά παρουσιάζει έκθεσή της ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι πάλι ένα ζήτημα, 8η αίτηση της Ελλάδας στο ταμείο αυτό και 5η όσον αφορά ε, το λιανικό εμπόριο. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ύφεση, μεγάλος ανταγωνισμός ε, που πλήττει εντός ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την Ελλάδα. Έχει μειωθεί κατά 63% το λιανικό εμπόριο από το 2008 και το 2016. 9 επιχειρήσεις αφορά 125 απολύσεις και 4,7 εκατομμύρια ε, για τον προπολογισμό του Ταμείου. Πρέπει να σας ε, Ενθυμίσω ότι 87% των απολυθέντων έχουν πάνω από, είναι πάνω από 55 ετών. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες συνέπειες στη δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να ξαναβρούν δουλειά ή να συνεχίσουν στα βιοδρομία τους. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ε, διαφάνεια, ε, να χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια, σωστά μεταξύ ε, των εργοδοτών και των ανθρώπων που θα πρέπει να είναι οι αποδέκτες αυτών των ποσών. Ε, θα υπάρξει επίσης και υποστήριξη της δημιουργίας επιχειρήσεων. Σας υπενθυμίζω ότι ε, οι συνεταιρισμοί μπορούν να είναι εναλλακτικές μορφές επιχειρήσεων που ανθίστανται περισσότερο στην κρίση. Ε, βεβαίως ε, ανταποκρίνεται σε μια επίγουσα κατάσταση η αίτηση αυτή. Είναι πολύ ε, απαραίτητο λοιπόν να δοθούν τα ποσά αυτά. Να τονίσω επίσης ότι ε, καλό θα ήταν ε, να σκεφτούμε μια συνεκτική στρατηγική εκ των προτέρων, να υπάρχει μια βιομηχανική προοπτική και μια δημοσιονομική προοπτική για να υπάρξει μια σχέση με τους τοπικούς μηχανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Μήπως υπάρχουν σχόλια? Όχι. Ευχαριστώ. πολύ. Εφόσον κανεί δεν ζητά το λόγο και σα έπεισε η παρουσίαση της εισηγήτρια, προθεσμία αποβολή τροπολογιών ε, μέχρι τις 3 το απόγευμα στις 10 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 20 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας και ε, θα υποβληθεί η γνωμοδότηση αυτή ε, στην μήνυ ολομέλεια των Βρυξελών ε, εδώ στο Νοέμβριο. Ο λόγος τώρα στον Τιέμο Βόλκεν για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω σύντομα κάτι για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Βρίσκω την πρόταση σωστή, βρίσκω και τον προσανατολισμό της ε, νομοθετικής πρότασης να δώσει δηλαδή στόχους στους νέους ανθρώπους στην Ένωση για Εθελοντισμό κλπ. Πραγματικά ιδιαίτερα ε, χρήσιμα και θετικά. Η πρόταση προβλέπει η χρηματοδότηση για το σώμα από το 2018 έως το 2020 να καταβληθεί κατά 75% από μεταφορές πιστώσεων, από ανακατανομές πιστώσεων και ιδίως από τα εξής προγράμματα Erasmus ΣΥΝ, από το πρόγραμμα για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, από αντιμετωπίσεις θεομηνιών, από το πρόγραμμα LIFE, από το Γεωργικό Ταμείο και από το Ταμείο ανάπτυξη της υπαίθρου και μόνο 25% θα είναι νοπό χρήμα. Η γραμμή της πολιτικής μου ομάδας αλλά και η γραμμή της Επιτροπής Προϋπολογισμών με οδηγούν να προτείνω ωστόσο μια άλλη γραμμή. Νέο πρόγραμμα, νέα χρηματοδότηση. Αυτά τα έχουμε πει και έχουμε εγκρίνει ήδη. Μετά από την υποβολή ωστόσο της γνωμοδοτήσεώς μου είχα την ευκαιρία να συζητήσω με συναδέλφους και να λάβω και άλλες λεπτομερείς πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θα επανεξετάσω την έκθεσή μου σε ό,τι αφορά την μεταφορά πιστώσεων από το πρόγραμμα Erasmus Συν, διότι μου κατέστησε σαφές ότι τα χρήματα που θα ληφθούν από το Erasmus Συν αντιστοιχούν στο τμήμα εκείνο το οποίο ε, διατίθεται για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών και ειδικά για τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή το Σώμα Αλληλεγγύης θα αναλάβει και τις δραστηριότητες των εθελοντών, θεωρώ ότι η μεταφορά αυτή πιστώσεων είναι τελικώς αποδεκτή. Αυτό όμως ισχύει μονάχα για αυτήν την μεταφορά πιστώσεων από το πρόγραμμα Ερασμοσύν. Δεν θα πρέπει να <clears throat> αγγιχθούν ωστόσο τα άλλα προγράμματα και θα πρέπει να ισχύσει η αρχή νέο πρόγραμμα, δηλαδή σώμα λίγη, νέα χρηματοδότηση. Θα προσαρμόσω την εκθεσή μου και βεβαίως ισχύει η 14η Νοεμβρίου ως προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Ευχαριστώ ε, κύριε Σιγητά. Από τους σκιώδεις ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Φερνάντες απουσιάζει. Ο κύριος Ντεπρέ. Ναι, Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τον εισηγητή μας. Όμως έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα η επιχειρηματολογία το δεν με Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα που θα το ε, γενιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λέμε διαρκώς ότι αυτό ήταν απόλυτη προτεραιότητα για μας. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν στο όνομα ποιας λογικής θα πάρουμε τα κονδύλια του Erasmus για να χρηματοδοτήσουμε αυτό το πρόγραμμα διαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου και είχαμε πει ότι ήταν πολύ ωραίο πρόγραμμα και ότι θα κοιτάξουμε να αποκτήσουμε τα πρόσθετα μέσα που χρειάζονται για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα και το καθεξής. Καταλαβαίνω την πνευματολογία του εισηγητού αλλά ε, επί της αρχής ενώ είναι σωστή δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να πάμε και να πάρουμε κονδύλια από ένα στρατηγικό πρόγραμμα όπως το θεωρούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσουμε ένα νέο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα δεν μπορώ να ε, λάβω τελική απόφαση πριν δω ποια θα είναι η τελική εκβάση του τριμερούς διαλόγου που θα οργανωθεί. Εγώ θα έλεγα η αντιπροσωπεία μας να ζητήσει να χρηματοδοτηθούν αυτό το πρόγραμμα από νέα κονδύλια. Ευχαριστούμε κύριε ε, Ντεπρέ, κύριε Κέλμελ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα σας ζητήσω συγγνώμη διότι δυστυχώς είχα άλλη ενηλυμένη υποχρέωση και προσήλθα με κάποια καθυστέρηση. Πράγματι, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ντεπρέ. Καταρχήν, το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι καλό είναι θετικό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όμως για τη χρηματοδότηση θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Συνολικά, για μένα είναι κάπως αδιαφανές από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια. Διότι αφενός λέμε ότι τα κονδύλια είναι απολύτω αναγκαία στι άλλε γραμμέ του προπολογισμού. Από την άλλη μεριά, όταν έρχονται νέε προτάσει, ψάχνουμε να βγούμε από εδώ και από εκεί για να πάρουμε, να κάνουμε μεταφορέ πιστώσεων. Ποια πράγματα ωστόσο έχουν προτεραιότητα οι προτεραιότητε πρέπει να γίνονται σεβαστέ και οι προτεραιότητε θα πρέπει αυτέ να καθοδηγούν το που διαθέτουμε τα χρήματα. Η κυρία Μπιού τη ενωτική αριστερά, όχι δεν έχετε πανέμβαση. Ο κύριο Τάραντ απεχώρησε. Η ευθυντή ποιο είναι εδώ εκ, εκ της ομάδος αυτής. Ποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ε, όχι, εσείς πάλι κύριε Ντεπρέ, όχι. Ορίστε εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομο σχόλιο. Εάν παίρνουμε χρήματα από ένα τμήμα του πιδελταπή για άλλη γραμμή. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί κατά τη γνώμη μου εάν μεταφέρουμε και δραστηριότητα από ένα τμήμα του προϋπολογισμού σε άλλο. Άρα πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά για το ποιες είναι οι δραστηριότητες που προτείνει το πρόγραμμα αυτό. Σε οποιοδήποτε οργανισμό που έχει προπολογισμό είτε πρόκειται την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε πρόκειται για ένα δημοτικό συμβούλιο, αυτό κάνει ο κόσμος. Όμως, εάν θέλουμε ανακατανομή, χωρίς να ακολουθούν οι δραστηριότητες, τότε θα πρέπει να αντισταθούμε στην πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχουμε λοιπόν νέα προγράμματα τα οποία εισέρχονται σε αυτή την φάση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και δεν προσελκύουν κατάλληλη νέα χρηματοδότηση, τότε ίσως είναι καλύτερα να περιμένουν τα προγράμματα αυτά μέχρι να συζητηθεί το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, αντί να παράγουμε μια σειρά από προγράμματα τα οποία θα είναι αποδυναμωμένα και όχι επαρκώς αποτελεσματικά. Καμιά φορά είναι καλύτερα να κάνει κανείς λιγότερα πράγματα, αλλά με καλύτερο τρόπο, παρά να κάνει περισσότερα πράγματα και να τα ποτίζει με το ποτιστήρι. Κατά τα άλλα συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Βέλκεν στην παρουσίαση τη εκθέσεώ του. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Βεβαίως και τις τροπολογίες θα καταδεχθούν. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε. Κύριε Ουρέλ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να αποσαφενιστούν κάποια στοιχεία για να απαντήσουμε στα σχόλια των βουλευτών. Πρώτα απ' όλα για την επαναδιάθεση κονδυλίων του Εράσμους. Να είναι σαφές ότι 100% της προτινόμενης επαναδιάθεσης προέρχεται από κονδύλια που αυτή τη στιγμή προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών. Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μάλλον Εθελοντών. Αυτές οι δραστηριότητες θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει παραμικρή επίπτωση για τις βασικές δραστηριότητες του Εράσμους, για την ότατη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ε, εκπαίδευση. Αυτό είναι μια βασική πτυχή της προτάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα αγγίξουμε τη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης, ούτε την επαγγελματική κατάρτιση, ούτε την εκπαίδευση. Αυτά όλα προβλέπονται από τα κονδύλια που ε, θα πήγαιναν στην υπηρεσία εθελοντών, που θα καλύπτονται πλέον από το σώμα αλληλεγγύης. Για τις υπόλοιπες δραμές, Η δική μας κατανόηση είναι ότι η πρότασή μας συνάδει πλήρως με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 6 Απριλίου φέτος όπου είχε καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει να χρησιμοποιηθούν ορθολογικά οι δραστηριότητες αυτές στα προγράμματα live λόγου χάρη και να υπάρχει ενιαίος συντονισμός. Βάσει λοιπόν και του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου κάναμε τη σχετική πρόταση. Ευχαριστώ να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις, αν χρειάζεται. Ευχαριστούμε κύριε Ουρέλ. Για τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών μιλάτε εσείς όμως. Ο κύριος Φράνς από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού. Καλημέρα σας. Θα συμφωνήσω με όσα είπε ο κ. Σουρέλ από τη Γενική Διεύθυνση Μπούτζ. Καμιά άλλη δραστηριότητα του Εράσμου ΣΥΝ δεν έχει επηρεαστεί από αυτή την επαναδιάθεση. Μάλιστα με την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μια ενιαία θηρίδα για την οργάνωση των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Στόχος των προγραμμάτων που συμβάλλουν στον ίδιο σκοπό δεν παραβιάζονται από το στόχο του σώματος αλληλεγγύης ίσα ίσα που βρίσκονται σε παράλληλη πορεία με τους στόχους αυτού του προγράμματος και αλληλοσυμπληρούνται. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η εθελοντική υπηρεσία η οποία αλλάζει σχήμα και φύση. Σωστά, κύριε Ντεπρέ. Ακριβώς, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι δέχομαι τη λογική του κυρίου Ρέλ, αρκεί να αποδείξουμε ότι τα μέσα που κινητοποιούνται τώρα για την εθελοντική υπηρεσία και ότι αυτά που θα χρειαστούν αύριο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι το ίδιο επίπεδου. Ωστόσο, η δική μου αποτίμηση και ίσως να ασφάλω είναι ότι τα χρηματοδοτικά μέσα για την εθελοντική υπηρεσία αυτή τη στιγμή είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση με τις ανάγκες που πρόκειται να προβλεφθούν και να αποδοθούν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οπότε, ε, πείτε μου κύριε Ουρέλ, ε, κάνω λάθος. Δεν χρησιμοποιούνται τόσες πολλές πιστώσεις από την υπηρεσία εθελοντών. Αύριο όμω θα υπάρξει κάποια διεύρυνση αυτών των δραστηριοτήτων στο επίπεδο του σώματο αλληλεγγύη. Δεν θα χρειαστεί αύξηση των κονδυλίων. Κάνω λάθο. Εγώ ήθελα να επιμείνω στο διότι φέτος γιορτάσαμε την 30 ετία του Εράσμους. Και τι δεν μας είπαν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι πραγματικά ε, έκαναν έναν εορτασμό ε, λυρικού χαρακτήρα, εγκομιαστικό. Και όταν μας είπαν τι είναι για τους πολίτες η Ευρώπη, ήταν το ευρώ και το Εράσμους. Το Εράσμος έχει προκαλέσει όμως ε, και απογοητεύσεις, γιατί μία στις δύο αιτήσει γίνεται δεκτή. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μην θέσουμε να αμφιβόλω τα μέσα του Εράσμους. Παρακαλώ κύριε Ουρέλ να καθησυχάσετε τον κύριο Ντεπρέ. Ευχαριστώ ευχαρίστως ε, πρόεδρε. Ο κύριος Ντεπρέ έχει δίκιο. Τα μέσα του Εράσμος για τις θελοντικέ δράσεις δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της νέας πρότασης. Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φρέσκο χρήμα. Προτείνει μία αύξηση των μέσων που προέρχονται από το Εράσμος και που δεν αρκούν. Βεβαιώνω βέβαια ωστόσο ότι το χρήμα που παίρνουμε από το Εράσμος δεν είναι άλλο από αυτό που θα απευθυνόταν σε ε, ε, εθελοντικές δράσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Τωμά, πολύ γρήγορα πρόεδρε. Εμένα αυτό που περισσότερο με ανησυχεί, γιατί όπως και εσείς θα σκέφτομαι, είναι ότι δεν είναι αρκετά τα κονδύλια του Εράσμους. Το Εράσμους το προβλέψαμε στην αρχή αυτού του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προσπαθώντας να το ε, επεκτείνουμε να το αυξήσουμε, διότι το Εράσμος είχε προκαλέσει απογοητεύσει. Είχε θεωρηθεί ένα κατεξοχήν εργαλείο που απευθυνόταν μόνο στην ε, πρώτη κατηγορία φοιτητών, στους καλύτερους. Η ζήτηση και η προσφορά λοιπόν ε, για το Εράσμος ε, συνεχίζονται, μεγαλώνουν Οπότε, ακόμη και αν καταλαβαίνω το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του οποίου όσα πήραμε από το Εράσμους ούτως ή άλλως αφορούσαν μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη, το πραγματικό ερώτημα είναι δεν έπρεπε τα μέσα αυτά να τα πάρουμε και να ενισχύσουμε το ίδιο το Εράσμος. Και για αυτό το νέο πρόγραμμα να χρησιμοποιηθούν νέα κονδύλια. Νέε δαπάνε, όπω είπε και ο εισηγητή, νέα έσοδα. Εδώ ναι, έχουμε νέε δαπάνε και δυστυχώ πάλι επαναδιάθεση. Άρα το ερώτημά μου είναι προστατεύουμε και επιτρέπουμε να μεγαλώσει και να διευρυνθεί η λειτουργία ενός προγράμματος που λειτουργεί τόσο καλά και, χρειαστεί, και χρειάζεται υποστήριξη. Ε, ευχαριστώ τους ΜΕΝ και τους ΔΕ για τα πολύ καλά σχόλια σας και τα επιχειρήματα που μας δώσατε εν ώψη του τριμερούς διαλόγου και την συνδιαλλαγή των προπολογισμών το 2018. Κύριε Ισηγητά, για να ολοκληρώσουμε. Πολύ σύντομα, <clears throat> κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τις και τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι ακριβώς αυτό που εξήγησε μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών μεταφέρονται ή πρόκειται να ή θα μεταφερθούν στο Σώμα Αλληλεγγύης, ακριβώς αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο του νέου προβληματισμού και γι' αυτό πρότεινα εγώ να διαγράψω το προηγούμενο περιεχόμενο μέρους της εκθεσεώς μου. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόγραμμα Εράσμος υποχρηματοδοτείται. Γνωρίζουμε επίσης όμως ότι το σώμα αλληλεγγύης είναι, ε, μάλλον το σώμα εθελοντών είναι μέρος του Έρασμος και τις δραστηριότητες του τώρα θα αναλάβει το σώμα αλληλεγγύης. Οπότε βρίσκω σωστό τα κονδύλια που δίνονταν πριν για το σώμα εθελοντών να μεταφερθούν τώρα στο σώμα αλληλεγγύης, το οποίο στην ουσία αποτελεί μια μετεξέλιξη της υπηρεσίας εθελοντών. Εν πάση περιπτώσει, ευχαρίστω θα αναλύσω τις τροπολογίες που θα μου υποβληθούν. Και ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Αρτουή. Θα πρέπει να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι το αργότερο στις 14 ενδεκάτου στις 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία στις 4 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, άλλωστε εκδίδουμε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Πολιτισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, και η οποία θα ψηφίσει την σχετική έκθεση τον επόμενο Ιανουάριο. Εσείς κύριε Κελμέλ ανταλλαγή πληροφοριών για εγκληματικότητα, για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους απάτριδες. Έχει το λόγο κύριε Κέλμελ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Με το Ευρωπαϊκό Ποινικό Μητρό για Επικούς Τρίτων Χωρών και Απάτριδες που ισχύει ήδη μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες οι χώρες μέλη για πρώην καταδίκες πολιτών τους. Είναι δυνατόν ως τώρα να γίνει μέσω ενός μηχανισμού hit, no hit, δηλαδή κάπως συμπτωματικού, δηλαδή μια διαδικασία hit, no hit σημαίνει ότι ρωτά κανείς, υποβάλλει την ερώτηση δηλαδή, και η απάντηση που λαμβάνει είναι αν υπάρχει πράγματι κάποιο στοιχείο στην τράπεζα δεδομένων ή όχι. Λίγο χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό για υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες και το γεγονό είναι <clears throat> ότι οι χώρες μέλη που ενδιαφέρονται για τέτοιες πληροφορίες σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να υποβάλουν ερώτηση σε όλες τις υπόλοιπε χώρες μέλη γιατί το σύστημα είναι αποκεντρωμένο. Επομένως, αν μια χώρα όπως η Γαλλία επιθυμεί να λάβει πληροφορίε για, μια, για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, πρέπει να υποβάλει σχετικό ερώτημα στις υπόλοιπε 27 χώρε μέλη. Βεβαίω πρόκειται για πολύ κοπιόδη και δαπανηρή υπόθεση και γι' αυτό το κόστος διαχείρισης της διαδικασίας αυτής ανέρχονται σε περίπου 78 εκατομμύρια ευρώ για όλε τι χώρε μέλη. Ε, Βεβαίω πρόκειται για ένα αποτρεπτικό νούμερο, αποτρεπτική διαδικασία του συστήματος αυτού που τα αρχικά του είναι εκρής. Πρόκειται τώρα εδώ για υπηκόους τρίτων χωρών και για απάτριδες. Το πρόβλημα δεν τίθεται για πολίτες των χωρών μελών, διότι βεβαίως αν θέλω να μάθω κάτι για κάποιον Ισπανό υπήκο, στέλνω μια ερώτηση στην Ισπανία. Για άλλους όμως υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μονάχα σε ένα 5% των περιπτώσεων. Και επειδή κατά τους πρόσφατους μήνες έχουν σημειωθεί οι γνωστές εξελίξεις και ιδίω λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων, καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαίο να γίνει μια ε, ε, συμπληρωματική νομοθετική πρόταση για να υπάρξει ένα κεντρικό, ένα συγκεντρωτικό σύστημα για την υποβολή ερωτήσεων και την άντληση δεδομένων. Η νέα πρόταση αναφέρεται σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα το οποίο θα ιδρυθεί από τον οργανισμό EU-LISA και αυτός άλλωστε το διαχειρίζεται όπου θα περιλαμβάνονται δεδομένα, δακτυλικά αποτυπώματα και ή δυνατόν και φωτογραφίες προσώπου των ε, προσώπων αυτών. Αυτό προσφέρει το πλεονέκτημα ότι θα επιτρέπει ευθεία πρόσβαση και για άλλους οργανισμούς, Eurojust, Europol, και βεβαίως καλύτερη ανταπόκριση της υποχρεώσεις που απορρέουν το καταστροφικό της Ιουλίσα για την χρήση τη Τράπεζα δεδομένων με πιο αποτελεσματικό τρόπο και για την δίωξη αλλά και για την πρόληψη των επιθέσεων. Με τη βοήθεια του συγκεντρωτικού αυτού συστήματο, οι χώρε μέλη θα μπορούν να διαπιστώνουν σε ποια άλλη χώρα μέλο ενδεχομένω υπάρχουν καταγραφέ στα ποινικά μητρώα σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα δεδομένα του συστήματος έκρης, ώστε ενδεχομένως να μπορούν να προλαμβάνουν τις θερμοκρατικές επιθέσεις ή πάντως να διαμορφώνουν αποτελεσματικότερα την δίωξη. Αυτό ισχύει βεβαίως και για όλες τις χώρες. Η νομοθετική πρόθεση στοχεύει στην κάλυψη κενών, ούτω ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα ε, σε πραγματικό χρόνο να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα σχετικά δεδομένα. Η χρηματοδότηση προβλέπεται ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το εφάπαξ κόστος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη και χρήση του συστήματος από το 2018 έως το 2020 σε 13 περίπου εκατομμύρια ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνεται το κόστος για την πρόσληψη πέντε ε, υπαλλήλων οι οποίοι θα εργαστούν ε, στην φάση ανάπτυξης του συστήματος. Το τρέχον κόστος για την ε, συντήρηση του συστήματος ανέρχεται σε 2,1 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το, άπαξ κόστος, το εφάπαξ κόστος για τις χώρες μέλη θα είναι της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος διαχείρισης θα ξεκινήσουν από 6 εκατομμύρια τον χρόνο όταν θα γίνεται πλήρης χρήση του συστήματος θα ανέρχεται πλέον σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Εάν τα συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά φτάνει σε ένα σύνολο της τάξης των 26 εκατομμυρίων ευρώ για, την, για το στήσιμο του συστήματος και τρέχοντα κόστη της τάξης των 17 εκατομμυρίων. Δεν είναι λίγα τα λεφτά αυτά, αλλά πρέπει να δούμε σαφώς ότι εάν δεν συμβεί αυτό τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα. Άρα εξοικονομούμε, διότι όπως είπα, το νυν ισχύον μη αποτελεσματικό σύστημα κοστίζει 78 εκατομμύρια το χρόνο. Αν βγάλουμε λοιπόν το κόστος που ανέφερα, μειώνουμε το κόστος διαχείρισης κατά 16 εκατομμύρια το χρόνο για το τρέχον κόστος διαχείρισης. Το κόστος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στα πλαίσια του προγράμματος για τη διάρκεια που προανέφερα μπορούν να καλυφθούν από τα κονδύλια του οργανισμού EU-LISA εάν ενισχύσουμε κατάλληλα τα κονδύλια. Και αυτό μπορεί να το καλύψει ο ισχύων δημοσιονομικός κανονισμός. Από το 2021 θα είναι μόνο το επαναλαμβανόμενο κόστος βέβαια για την διαχείριση του συστήματος, τη συντήρησή του δηλαδή ετησίως. Κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να καλύπτει το δικό της κόστος για την χρήση του έκρης. Θεωρώ λοιπόν την εκτίμηση κόστους για τον ευρωπαϊκό προϋπολισμό ως αναλογική και επαρκή. Παρόλο που το τίμημα για το νέο σύστημα και για τον ευρωπαϊκό προϋπολισμό και για τις χώρες μέλη είναι υψηλότερο από την πρόταση που είχε γίνει του 2016, οι σημαντικέ εξοικονομήσει που θα προκύψουν κατά την διαχείριση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και γι' αυτό το λόγο η διαδικασία στο σύνολό τη για μα είναι συμφέρουσα και ταυτόχρονα οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ποιότητας. Ζητώ ωστόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει στον οργανισμό η Ιουλίσα αλλά και στις χώρες μέλη ώστε κατά την καθίδρυση και διαχείριση του συστήματος και συντήρησή του να γίνει κάθε δυνατή εξοικονόμηση κόστους. Και αυτή θα είναι η γνωμοδότησή μας για την αρμόδια εξουσίας επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Κελμέλ για την παρουσίασή σας. Είναι προφανές ότι η προστιθέμενη αξία της προτάσεως είναι σημαντική. Κύριε Ντεπρέ, νομίζω ζήτησατε το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και απολύτως με αυτά που μόλις είπε ο συνάδελφος Κέλμελ, ε, η τροποποίηση λοιπόν που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου φαίνεται συνετή, ειδικότερα όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την ε, ε, επιπλέον λειτουργικότητα που δημιουργεί. Συμφωνώ επίσης με τον συνάδελφο ότι είναι λογικό το κόστος χρηματοδότησης και αναλογικό, δεν ξέρω ακριβώς τι όρους χρησιμοποιήσατε, δεν θυμάμαι πια, αλλά νομίζω ότι είναι λογική και αναλογική λογική αυτή η πρόταση. Θα ήθελα να ε, Στραφώ τώρα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια βελτίωση που θα μα δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τα, μηνικά, τα ποινικά μητρώα των ε, υπηκών τρίτων χωρών. Αυτή τη στιγμή η αναζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά πρέπει να μα χρησιμεύσει και σε κάτι. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή θα δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα το οποίο λέγεται ETIAS ε, που είναι η εκ των προτέρων άδεια για την είσοδο στην ε, Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Συνδέεται αυτό μεταξύ του νέου συστήματος ETIAS με το ΕΚΡΙΣ, γιατί μου φαίνεται ενδιαφέρον όταν φτιάχνουμε κάτι που έχει και ένα επιπλέον κόστο, τουλάχιστον η διαλειτουργικότητα, αν δηλαδή μας επιτρέπει το ΕΚΡΙΣ να, πούμε, να δούμε ποιο είναι το ποινικό μητρό των υπηκών τρίτων χωρών, νομίζω ότι αυτό έχει νόημα ε, να ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και το συνδέω αυτό και με το σύστημα των ε, της χορήγησης θεωρήσεων είναι και ένα επιχείρημα που αφορά τον προϋπολογισμό αυτή εφόσον θα υπάρξουν πιστώσεις υποχρεώσεων ο στόχος είναι να υπάρξει και ε, κέρδος από την επένδυσή μας ε, αυτή. Να, ε, θα είναι δύσκολο λοιπόν να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα χωρίς να αυξηθεί το κόστος. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν με το σύστημα VIS, το σύστημα για τις θεωρήσεις και το ETIAS είναι εξασφαλισμένη η κυρία Γουαρδία Θαβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτε παραπάνω. Νομίζω ότι το θέμα της διαλειτουργικότητας μετά από την ευελιξία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται περισσότερο στην Επιτροπή μας. Ε, το είπε και ο κύριος Ντεπρέ. δεν είναι το πρώτο θέμα επί του οποίου κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνούμε με την άποψη του κυρίου Κέρμελ, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι περίπλοκη, περίπλοκο το σύστημα, ε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια στον προϋπολογισμό προς αυτό. Συμφωνούμε λοιπόν ε, με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, θέλω πάρω το λόγο. Όχι. Κύριε Ιουρέλ, μήπω θέλετε να απαντήσετε στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις του εισηγητή και των συναδέλφων. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόλμελ για την υποστήριξη του ε, στην πρότασή μας και όλους τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους του που εξέφρασαν την υποστήριξη προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις τροποποιήσεις. Έχω ένα σχόλιο να κάνω αυτή τη στιγμή και που έχει να κάνει με την τροπολογία 4 αύξηση της συχνότητας αξιολόγησης. Εμείς θα προτιμούσαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αλλάξει η συχνότητα αξιολόγηση, να παραμείνει στα τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργία του συστήματο και κάθε τέσσερα χρόνια μετά. Ε, γιατί, γιατί υπάρχουν ήδη εκθέσεις ε, οι οποίες προβλέπονται από τον οργανισμό e και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι είναι επαρκή, επαρκής αυτές οι εκθέσεις για να παρέχουν πληροφορίες σε σχέση με το σύστημα. Για το ερώτημα τώρα του κυρίου Ντεπχέ, ε, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό το ερώτημά σας και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν, έβγαλα, δεν, δεν βρήκα πληροφορίες σχετικά, σχετικά στην ε, ενημέρωση. Θα το διερευνήσω και θα σας απαντήσω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μάλιστα. Η διαλειτουργικότητα είναι μια ε, αιμονή ε, ε, μα, η οποία πρέπει να τη δώσουμε σάρκα και οστά. Το λόγο λαμβάνει πάρα ο κύριο Κιόλμελ. Ευχαριστώ και εσά, κύριε Πρόεδρε και του συναδέλφους μου καθώς και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις του. Αναμένω με ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες. Θα εξετάσω και πάλι αυτές που έχω ήδη λάβει, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν. Τίνω για την ώρα ότι να, να, να, να ε, θεωρήσω ότι η περίοδη αξιολογήσεως που ε, προβλέπονται ήδη είναι επαρκής. Θα χρειαστεί να υποβάλλονται και εκθέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει έξτρα εργασία, διότι αξιολόγηση είναι αξιολόγηση. Και εάν επεκταθεί και σε άλλους τομείς, παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το σύστημα έκρηση. Θα τα κοιτάξω πάντως. Ευχαριστώ και πάλι πολύ και ευχαριστώ για την υποστήριξη που προσφέρουν οι συνάδελφοι στην πρότασή μου. Ο πρόεδρος Αρτουή. Ευχαριστώ κύριε Κέρμελ. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου τη 12η Μεσημβρινή, 4 Δεκεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, η ΔΕ Αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, 24 Ιανουαρίου. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Έχετε ε, θέματα στα διάφορα. Δεν βλέπω κανένα. Η επόμενη συνάντησή μας ε, θα λάβει χώρα στις 22 και σίγουρα και στις 23 Νοεμβρίου. Λίγη συνεδρίαση.